τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Ενημερώνω τα μέλη για τα εξής. Στη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου του 2019, οι συντονιστές ε, της Επιτροπής Αναφορών ενέκριναν το σχέδιο μερίσας διάταξης ε, για τη συνεδρίαση της 4ης και 5ης ε, Σεπτεμβρίου, αυτή που έχουμε τώρα δηλαδή. Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Αναφορών θα οργανώσει μία ακρόαση για τη ΦΑΤΚΑ με τη συμμετοχή των αναφερόντων, των κρατών μελών και ενός εκπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΕΚΟΝ, εάν οι Επιτροπές αυτές το επιθυμούν. Επιπλέον, ε, ορίστηκε ο εισηγητής για την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του 2018. Ε, αναλαμβάνει ένας εισηγητής από το ΕΛΚ και ο... είναι ο κύριος Πίτερ Γιάρ. Επίσης, αποφασίστηκε η σύσταση του δικτύου αναφορών, το Petition Network, και να ζητήσουμε από όλες τις υπόλοιπες επιτροπές, αυτή τη στιγμή συσταθούν σε σώμα, να ορίσουν τουλάχιστον ένα ευρωβουλευτή, στο μέτρο του δυνατόν κάποιον ο οποίος να μην είναι μέλος της Επιτροπής Αναφορών. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, σημείο 5, που είναι η παρουσίαση Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία τη με την Επιτροπή Αναφορών. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο φυσικός ε, ε, συνομιλητή τη Επιτροπής Αναφορών όταν διαβιβάζονται οι αναφορές, ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την τήρηση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Να καλωσορίσω εδώ τον Ερίκο Φόρτη, Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση των Διοργανικών Σχέσεων τη Γενική Γραμματεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Φόρτη, λοιπόν, έχει το λόγο για 10 λεπτά. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Καταρχάς, ε, να σας συγχαρώ για το αποτέλεσμα της εκλογής σας εδώ ως Προέδρου αυτής της Επιτροπής. Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει στη νέα Επιτροπή Αναφορών. Για μας φυσικά στην ε, Επιτροπή και στο Γενικό Γραμματέα ε, η Επιτροπή αυτή έχει μεγάλη σημασία. Είναι η φυσική προστασία των ε, δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κανάλι άμεσης επικοινωνίας με το Κοινοβούλιο. Είχαμε ως τώρα εξαιρετική συνεργασία με την Επιτροπή σας την τελευταία νομοθετική περίοδο. Είχαμε διαρθρωτικό διάλογο με τον Αντιπρόεδρο και όλη την Επιτροπή. Επίσης είχαμε μια πολύ καλή σχέση, φιλική σχέση με την ομάδα σας και τονίζω και δίνω έμφαση στην ανάγκη να συνεχίσει αυτή η πορεία, αυτή η εμπειρία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τις ανησυχίες ε, που βαρύνουν ε, τους πολίτες μας. Επίσης, θα μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα μη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας μη σωστή εφαρμογή τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιτροπή σα είναι συμπληρωματικό στοιχείο. Ε, είναι πολλέ φορέ το έναυσμα που μας οθεί στο να βρούμε τις περιπτώσεις κακής εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα και αδειμονούμε, ε, ανυπομονούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί σας. Η συνεργασία μας έχει τρία επίπεδα. Πρώτον, έχουμε το πολιτικό επίπεδο. Ο διαρθρωτικός διάλογος με τον Αντιπρόεδρο της ε, τωρινής και της μελλοντικής, ελπίζω, Επιτροπής. Σύντομα. Μετά έχουμε την καθημερινή συνεργασία της ομάδας μου με την ομάδα σας. Και έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό, την ετήσια έκθεση για τις αναφορές προτείνω σε αιτήσια βάση, χωρίς να ξέρουμε βέβαια ε, και άλλη, την πιθανότητα να υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Ε, γι' αυτό δεσμεύομαι προσωπικά. Επίσης, παρόλο που έχουμε μια καλή συνεργασία, υπάρχουν ακόμα θέματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, επιδέχονται βελτίωσης αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί να εξετάσει όλα τα ζητήματα που τρέχουν. Πρέπει να μάθετε και θέματα ουσίας βέβαια, αλλά ένα από τα σημαντικά ζητήματα είναι οι προθεσμίες. Έχουμε επί της αρχής τρεις μήνες για να απαντήσουμε σε μία αναφορά. Βέβαια, στην εποχή του ίντερνετ οι τρεις μήνες φαντάζουν δεκαετίες. Κάποιες φορές είναι αδικαιολόγητο γιατί κάποια αναφορά μπορεί να είναι επίγουσα, η ανησυχία του πολίτη να είναι επίγουσα. Υπάρχουν όμως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις Υπάρχει περισσότερη ανάγκη να τηρηθεί αυτό το τρίμηνο, γιατί μπορεί να έχουμε ένα περίπλοκο ζήτημα, όπου ε, πλέκονται λίγο τα όρια μεταξύ της εθνικής αρμοδιότητας και της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διερευνηθεί ένα θέμα. Επίσης, είναι σημαντικό ε, γιατί ε, σε μία αναφορά η Κομισιόν δεν απαντά σε διοικητικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο ε, κολεγίου των επιτρόπων. Είναι μια γραπτή διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Βέβαια, προσπαθούμε λίγο να βρίσκουμε μια πιο απλή λύση σε κάποια στάδια της διαδικασίας. Πολλές φορές, ας πούμε, αν έχουμε μια αναφορά ε, σε μια γλώσσα και πρέπει να περιμένουμε την μετάφραση, ενδεχομένως, αν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πρακτικό, πιο πραγματιστικό τρόπο να κερδίσουμε χρόνο. Επίσης, πρέπει να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής που διαθέτουμε. Αναγνωρίζω ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση των εργαλείων μας, να είναι πιο να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους και γενικά να είναι πιο αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα με την ομάδα σας τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Η διοικητική λοιπόν διαχείριση είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η σχέση μεταξύ του υποκειμένου της αναφοράς και της παράβασης. Έχουμε ένα σύστημα βάσει του οποίου οι διαδικασίες επί παραβάση που σχετίζονται με μία αναφορά μπαίνουν μπροστά της και αυτό πρέπει να το δουλέψουμε λίγο. Φυσικά από την Επιτροπή σας μπορούμε να έχουμε ε, κάποια ε, ενημέρωση εμείς ως Κομισιόν για τα στοιχεία της νομοθεσίας ε, που δεν λειτουργούν σωστά. Όμως δεν είναι ότι και όλες οι αναφορές οδηγούν σε τέτοια θέματα. Δεν είναι πάντοτε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Πολλές φορές δεν εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο. Κάποιες φορές επίσης ε, μέσα από μια πιλωτική διαδικασία ή προηγούμενη διαδικασία επί παραβάση, η Κομισιόν έχει ήδη εξετάσει μια αναφορά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε το περιβάλλον, την εσωτερική αγωνά, την υγεία, την ενέργεια, τις, μεταφοράς, τις μεταφορές και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Για το περιβάλλον έχουμε περίπου, είχαμε περίπου 200 αναφορές το 2018, τις οποίες απαντήσαμε. Πολλές φορές είχαμε και πολλές απαντήσεις για την ίδια αναφορά τις αναφορές το 40% ήδη είναι υποδιαρεύνηση. Μιλάω για το ζήτημα το οποίο έχει γύρει ο αναφέρον. Έχω ε, ματερές, ε, ε, επεξεργασία λιμάτων, ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις επίσης που ένα κομμάτι της αναφοράς σχετίζεται με έρευνα που ήδη διεξάγεται. Άρα, αν βελτιώσουμε την επικοινωνία, αν υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, θα έχουμε αποτελέσματα. Έχω δει πολλές εκθέσεις από την Επιτροπή Αναφορών. Ε, θέλετε περισσότερη πληροφόρηση για τις διαδικασίες επί παραβάση. Πού βρισκόμαστε για να μπορέσετε και να αξιολογήσετε καλύτερα αν μία αναφορά έχει να κάνει με ένα καινούριο ζήτημα ή με ένα που ήδη τρέχει. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια μπορούμε να βρούμε προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται μέσω της διαδικασίας επί παραβάση και να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία ή να βρούμε θέματα που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Καλό είναι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να ενημερώνουμε τους αναφέροντες. Επειδή η Επιτροπή σας έρχεται και σε επαφή με τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, έχουμε ήδη ξεκινήσει με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ε, σε διοικητικό επίπεδο μία προσπάθεια να αξιολογήσουμε κατά πόσο η έρευνα γίνεται με σωστή βάση. Δεν αποφασίζουμε τίποτα, απλώς δίνουμε ε, τα γεγονότα τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζονται οι υπηρεσίες του Ombudsman για να ε, δουν εάν ε, η έρευνα γίνεται επί της σωστής βάσεως. Επίσης παρατήρησα ότι ο ρόλος της Κομισιόν είναι κρίσιμος ως προς την παροχή βοήθειας προς τους αναφέροντες να βρουν διέξοδο. Αν είναι κάτι εντός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τον αναφέροντα να ε, βρει δικαίωση ε, απέναντι στις εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα να θίξω λίγο πολύ. Υπάρχουν και κάποια άλλα, ε, όπως ας πούμε οι ορφανές ή οι λανθάνουσες αναφορές όπως τις λέτε εσείς. Εκεί μπορεί να γίνει περισσότερη δουλειά. Να συνοψίσω, κυρία Πρόεδρε, σύντομα λοιπόν το μήνυμά μου προς εσάς και προς τα μέλη της Επιτροπής σας. Θα εργαστούμε επί του χρόνου απάντησης από την πλευρά της Κομισιόν, αντίδρασης από την πλευρά της Κομισιόν. Θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία για τις ε, διαδικασίες επί παραβάση. Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των λανθανουσών αναφορών. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα που θέλω να σας δώσω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φόρτη, και για την πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση και τις εξηγήσεις που μας δώσατε και εμείς προσβλέπουμε στη μεταξύ μας συνεργασία ώστε να βελτιώσουμε τη διαδικασία και να έχουμε και γρήγορες απαντήσεις. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θα έχουν, θα το λόγο. Κύριε Άουκεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά, με μεγάλη χαρά ακούσαμε ότι θα προσπαθήσετε να επιταχύνετε Εμείς ε, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ευαισθητοποίηση. Και όταν έρχεται κάποιος ε, σε εμά, ε, τους λέω ότι είναι καλό και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι το εκτιμάτε κι εσείς. Όμως μετά υπάρχουν κάποιες εσωτερικές, κάποια προβλήματα εσωτερικά. Η Κομισιόν πρέπει να είναι θεματοφύλακα στις συνθήκες για την τήρηση της νομοθεσίας. Εκεί όμως ε, το ρόλο αυτό πρέπει να πω δεν τον έχετε εκπληρώσει απόλυτα. Το να έχετε καλές διμερείς επαφές ε, δεν είναι το παν. Το παν είναι να είναι σαφές ότι η νομοθεσία λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες για ορισμένες οδηγίες που έχουν να κάνουν τη φύση, για παράδειγμα. Και η Επιτροπή ΕΜΒΗ με ομοφωνία και αυστηρότητα είχε ζητήσει από την Κομισιόν να είναι έξω από το ΡΕΦΤ, για παράδειγμα, ε, η συγκεκριμένη νομοθεσία για τη φύση. Η νομοθεσία είναι καλή και δεν είναι το πρόβλημα η ποιότητα, αλλά η εφαρμογή. Δεν εφαρμόζονται δηλαδή τα νομοθετήματα και εδώ είναι δική σας δουλειά. Πρέπει να δραστηριοποιηθείτε πολύ περισσότερο και ελπίζω και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αντιληφθεί. Αν θέλουμε να είναι αξιόπιστη ένωση και η νομοθεσία μας πρέπει να φροντίζουμε όταν ο νόμος ε, περνάει να είναι νόμος, να εφαρμόζεται δηλαδή στα κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν οι αναφορές αφορούν μη τήρηση νομοθεσίας ε, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται και θα έπρεπε να είναι και λιγότερες ουσιαστικά και θα ήταν λιγότερες αυτές οι αναφορές αν η Κομισιόν έκανε πιο σωστά τη δουλειά της. Ή κάποιες φορές καθυστερεί πάρα πολύ η διεκπαιρέωση, η συζήτηση επί μιας αναφοράς και δεν ε, είναι και αυτό σωστό. Άρα δεν θα έπρεπε να βασίσετε τόσο πολύ στην Επιτροπή Αναφορέ, αν τη χρειάζεστε τόσο πολύ την Επιτροπή Αναφορέ και τι αναφορέ, αλλά έπρεπε να κάνετε εσεί πιο πολλά πράγματα. Κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν. Είναι σπάνιο να έρχεται κάποιος και να λέει ότι δεν μιλάμε για αυτά τα οποία ε, πηγαίνουν καλά, δηλαδή να μιλάμε για μισή ώρα ε, και να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά ε, ξεκινάμε λέγοντας τι δεν πάει καλά και τι μπορεί να βελτιωθεί. Από αυτή τη βάση νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε πολύ καλά, μπορούμε να συμφωνήσουμε και με το ότι είπατε για την τρίμηνη προθεσμία που δύσκολα τηρείται και πράγματι είναι αναγκαίο να δίνονται πιο γρήγορα απαντήσεις. Μήπως να αλλάξω μικρόφωνο γιατί κάπως περίεργα ακούγεται. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται η ε, συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αναφορών. Δεν ξέρω τι φταίει με τα μικρόφωνα. Irgendeiner hat die Rückkopplung. Ähm, zwei Fragen. Δύο ερωτήσει. Η διαδικασία παραβάση, η παράβαση της νομοθεσίας είναι αυτό που μας αφορά και είναι ένα θέμα που αφορά γενικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε πιο γρήγορη αντίδραση. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε όμως όταν πρέπει μια αναφορά και όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για κάποια κατασκευαστικά και είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Εμείς ως Επιτροπή δεν έχουμε λόγο να διορθώσουμε τη συμπεριφορά των κρατών μελών σε αυτή τη φάση του σχεδιασμού. Όταν όμως βέβαια έχει αναγερθεί κάτι, είναι δύσκολο να διορθωθεί η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να το βλέπουμε αυτό. Να βλέπουμε αν έχουμε μια αναφάση φάση του σχεδιασμού, είναι δυνατόν και εκεί να μπορούμε να δράσουμε πιο αποφασιστικά. Και μια παρότρινση. Το είπατε κι εσείς. Πρέπει με ειλικρίνεια να βλέπουμε πού είμαστε αρμόδιοι και πού δεν είμαστε αρμόδιοι. Το είπατε κι εσείς. Υπάρχουν κάποιες ε, και για μας δύσκολες αναφορές ε, που πραγματικά ε, μας λυπεί πάρα πολύ ε, το γεγονός ότι είμαστε όμως αναρμόδιοι για κάποια θέματα πάρα πολύ προσφυλή για εμάς ή σημαντικά. Δεν ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν, να δούμε τι συμφωνία θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον. Πάντω η δική σας ομιλία μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ξεκινήσατε με τα θέματα όχι που είναι ήδη καλά, αλλά με αυτά που μπορούμε να βελτιωθούν περισσότερο. Ευχαριστώ. Ε, very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση στην αρχή αυτού του Κοινοβουλίου ε, για τις σχέσεις με την Κομισιόν. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρξει πολύ κριτική από την Επιτροπή μας για το τι είπε η δική σας πλευρά σχετικά με μια αναφορά ή όχι. Όμως, ε, για να ξεκινήσουμε επικοδομητικά, ας δούμε τα καλύτερα παραδείγματα από τα τελευταία χρόνια όπου είχαμε καλή συνεργασία με διάφορους γενικούς διευθυντές της Επιτροπής ε, και με την Επιτροπή Αναφορών και ας μιλήσουμε για τις λύσεις που βρέθηκαν. Όπως είπε και η Μάργαρετ, εμείς χρειαζόμαστε στο Κοινοβούλιο μια κομισιόν η οποία θα είναι εκεί, θα κρατά τη θέση της στεναρά ως θεματοφύλακας των συνθήκων, έτσι ώστε οι πολίτες να δικαιώνονται και να μην χρειάζεται να περνάει πολύς χρόνος τρεις μήνες για να αναλυθεί μία αναφορά ε, είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε υπό το πρίσμα των πολλών ετών που χρειάζονται πολλές φορές να περάσουν ε, στην διαδικασία επί παραβάση. Ε, όταν ζητάμε από ένα κράτος να επανορθώσει και μετά από πέντε χρόνια πάλι κάτι δεν γίνεται και επανέρχεται η αναφορά και περνάνε 10 και 15 χρόνια ε, για ένα θέμα όπου όλοι είχαμε συμφωνήσει ότι υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και δεν έχει ληφθεί δράση από το κράτος μέλος για να επανορθώσει, καταλαβαίνετε. Αναγνωρίζω ε, την χρονική πίεση. Για τους πολίτες η Ευρώπη πολύ συχνά κινείται πολύ, πολύ αργά. Καλό είναι λοιπόν οι πολίτες να παίρνουν όσο πιο γρήγορη απάντηση μπορούν όταν λαμβάνουμε μία αναφορά, γιατί εμείς μπορούμε να εξηγήσουμε μεν τα άτομα στην εκλογική μας περιφέρεια, στους φίλους μας, γιατί μια διαδικασία αργει Όμως η απάντησή μας προς αυτούς ας είναι γρήγορη για να καταλάβουν ότι του λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Τρεις μήνες πολλές φορές είναι πολύ καιρός. Βλέπω ότι πολύ συχνά ζητάμε τη διαδικασία, την έκτακτη διαδικασία ε, για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, ε, από την ε, θετική πλευρά να δούμε λίγο τα πράγματα. Καλό είναι να δίνουμε κάποια παραδείγματα στους νέους συναδέλφους, τα νέα μέλη της Επιτροπής, για να τους δώσουμε ένα κίνητρο Ας πούμε, η επισφαλής εργασία στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, αναφορές ε, σε αυτήν εδώ ε, την Επιτροπή με πολίτες που μιλάνε για συμβόλαια μηδέν ωρών και πριν από τις ευρωεκλογέ στο Στρασβούργο είχαμε την τελευταία μας μάχη για την ομοθεσία που είχε στόχο να βελτιώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο ε, υποφελείται από τη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και των ε, νομικών της ε, Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης. Επίσης, η ομάδα εργασίας για, για τα παιδιά. Αυτή ήταν μια δύσκολη ομάδα, όπως είπε και ο Πέτερ, έχουμε ευαίσθητα θέματα, όμως όταν εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εκπροσωπούμε τους πολίτες, να είμαστε φωνή τους τους θεσμούς, αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα ε, στα οποία το παραδεκτό ε, αμφισβητείται. Έχουμε περιπτώσεις που δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη οι παιδιά που εκλάπηκαν στην ε, Ισπανία και έπρεπε να βρούμε τα, τι γίνεται πηγαίνοντα στη Μαδρίτη. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία ε, με την ε, μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης που ασχολείται με τα δικαιώματα των θυμάτων. Αυτά είναι καλά παραδείγματα που πρέπει να τονίσουμε, να τα λέμε μεταξύ μας. Πού λειτουργεί καλά το πράγμα για να δείξουμε στα νέα μέλη μας τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Επιτροπή Αναφορών και πώς η καλή συνεργασία με τις επιτροπές πολιτικής του Κοινοβουλίου ε, φέρνει ε, συγκεκριμένη έκβαση, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Φόρτη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω σημειώσει αρκετά μηνύματα προς εμένα και θα απαντήσω πολύ γρήγορα για την τελευταία παρέμβαση της κυρίας Κίρτον ε, Ντάρλινγκ. Θεωρώ ότι είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ε, πού ε, έχουμε αποτελέσματα. Στην τελευταία θητεία έχουμε 700 συναδέλφους που τελικά είχαν την ευκαιρία να ε, επισκεφθούν την Επιτροπή σας και το καθήκον μου είναι να τους ενθαρρύνω να συνεργαστούν στενά μαζί σας για αυτές τις υποθέσεις. Συμφωνώ βεβαίως για το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι δεν ε, έχουμε μόνο τις αναφορές αλλά εφαρμόζεται και η νομοθεσία. Το μήνυμα θα διαβιβαστεί. Ε, σημειώνω ήδη ότι υπάρχει μείωση στον αριθμό των αναφορών τα τελευταία ένα-δυο χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά το μήνυμα θα διαβιβαστεί κυρίως ε, στα νέο μέλος ε, του Σώματος των Επιτρόπων που θα είναι αρμόδιος ε, για τα θέματα αυτά και θα ενημερωθεί. Θα είναι μεταξύ των στοιχείων που θα του γνωστοποιήσουμε. Τώρα, το θέμα που ανέφερε ο κύριος Γιάρ, ένα από τα καθήκοντά μας δεν είναι απλώς να απαντούμε στις αναφορές ε, και να ε, γίνονται σωστά τα πράγματα, αλλά επίσης να βοηθήσουμε και τους αναφέροντες ε, που ο μόνος τρόπος που έχουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους είναι να προσφύγουν στην Επιτροπή Αναφορών η οποία ίσως δεν έχει την κατάλληλη αρμοδιότητα, είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αναφέροντες ε, στο σωστό επίπεδο, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ε, και αυτό φυσικά είναι κάτι που θα κάνουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Φόρτη. Ζητώ συγγνώμη γιατί η κυρία Σδάνοκα είχε ζητήσει το λόγο, δεν την είδα. Κυρία Σδάνοκα, έχετε το λόγο. Ίσως ε, απλώς ε, για να συνεχίσω τις, ε, την ερώτηση που έθεσε ο κύριος Γιάρ. Αναφερθήκατε στα όρια των αρμοδιοτήτων και το κατά πόσον θα πρέπει να αποφασίσουμε αν εμπίπτει σε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι ε, μια αναφορά. Από την εμπειρία ε, που έχουμε εμείς στην Επιτροπή Αναφορών είναι ότι υπάρχει διαφορά στην προσέγγιση των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής μας και ε, εμείς θεωρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Η Επιτροπή όμως αποφασίζει ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Και πολλές από τις αναφορές, της ε, εκθέσεις μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λένε ότι το ΤΑΔΕ δεν εμπίπτει ε, στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. τέθηκε το εξή. Ε, υπήρχε για παράδειγμα ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκεί αμφισβητούνταν το κατά πόσον θα πρέπει να συζητηθεί, αλλά εμεί το κάναμε. Ε, θα ακούσουμε και την νομική υπηρεσία τώρα, ε, η οποία και αυτή εξέφρασε ανησυχίε για την προσέγγιση σα. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Και όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Στάνοκα, θα περάσουμε τώρα στο σημείο 6 που είναι η παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας ε, για τη συνεργασία της ε, με την Επιτροπή των Αναφορών και να καλωσορίσω την Μαρία Χωσέ Μαρτίνε Φιγκλέσιας, ε, Διευθύντρια του Τμήματος Νομοθετικών Θεμάτων της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μαρτίνε θα παρουσιάσει τι ακριβώς κάνει η νομική υπηρεσία και πώς υποστηρίζει την Επιτροπή μας. Θα εξηγήσει πώς και πότε γίνεται διαβούλευση με την νομική υπηρεσία και θα αναφερθεί επίσης και στην νομολογία που σχετίζεται με τις αναφορέ αναφορέ, το παραδοκτό των αναφορών και την παρακολούθησή τους. Να τις δώσω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσουμε την ομάδα μας και τη δουλειά μας στην Επιτροπή ε, τώρα στην αρχή της ε, θητείας. Πριν ε, κάνουμε την εισαγωγή στη νομική υπηρεσία να σας συστηθώ. Είμαι η Διευθύντρια Νομοθετικών Θεμάτων. Είναι Υπάρχει Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με τις αρμοδιότητες ε, όλων των επιτροπών για τις εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Ε, Εντό της Γενικής Διεύθυνσης, ε, το τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο για τις αναφορές είναι το τμήμα Δικαιοσύνη και Πολιτικών Ελευθεριών. Τμηματάρχη είναι ο κύριος Ντανιέλ Μπαρά, εδώ δίπλα μου, και ο νομικό ο οποίος ασχολείται καθημερινώς με την Επιτροπή Αναφορών, είναι ο κύριος Λιούκανεν, εδώ και αυτό. Και έχουν κάτι κοινό. Και οι δύο έχουν ε, υπάρξει δικαστές στις χώρες τους πριν ενταχθούν ε, στο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την περίπτωση ε, της ε, Επιτροπής μας το να υπάρχει τέτοια εμπειρογνωμοσύνη. πιστεύω ότι δύο λόγοι αιτιολογούν την ανάγκη για νομική συνδρομή και νομικές συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδίω μετά από την έναρξη ισχύω της συνθήκη της Λισαβόνα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πολιτικές και δραστηριότητες ε, και οι δραστηριότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει ε, να συλλαμβάνονται και να εφαρμόζονται εντό νομικού πλαισίου σεβόμενοι πλήρως τη συνθήκη και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της ε, παραπομπής, η οποία ισχύει ε, για τα ευρωπαϊκά όργανα ως εξής. Σημαίνει ότι κάθε ευρωπαϊκό όργανο, διαβάζω το άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε ευρωπαϊκό όργανο θα πρέπει να δρά εντός των ορίων των εξουσιών που του εκχωρούνται από τις συνθήκες και βάσει τις διαδικασίες, ε, τους όρους και τους στόχους που τίθενται. Η βασική αποστολή λοιπόν της νομικής υπηρεσίας είναι να συνδράμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σέβεται αυτές τις αρχές και κατά αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει για την ασφάλεια δικαίου της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την περίπτωση εσείς έχετε μια συγκεκριμένη αναφορά εσείς ως, ε, ε, αποστολή, συγγνώμη, εσείς ως Επιτροπή Αναφορών, διότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα, ε, είναι εγγεγραμμένο στις συνθήκες και ε, η δική σας αρμοδιότητα είναι να εφαρμόζετε αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα, την άσκηση αυτού του δικαιώματος που συνδέεται στενά με τις βασικές αξίες της έννοιας, όπως, της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της συνθήκης το νομικό στοιχείο στη δουλειά σας, ε, στην ουσία ε, περιορίζεται στα κριτήρια για το παραδεκτό μιας αναφοράς, που είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να ε, επανεξετάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και εδώ η βασική δουλειά της νομικής υπηρεσίας είναι να σας βοηθήσει στον τομέα αυτό, να σας βοηθήσει να καθορίσετε σε αυτό το στάδιο του παραδεκτού ή μη, κατά πόσον ένα θέμα, ε, το αντικείμενο της αναφοράς, εμπίπτει στην ευρωπαϊκή δραστηριότητα και ε, αφορά ε, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παραδεκτό είναι διτό. Υπάρχει ο νομικός κίνδυνος, ο οποίος αφορά την απόφαση να θεωρηθεί παραδεκτή μια αναφορά ε, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί και να θεωρηθεί μη παραδεκτή. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει άποψη ότι το νομικό πρόσκομα επιλύεται εάν μία αναφορά θεωρηθεί παραδεκτή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, ελοχεύει ο ίδιος κίνδυνος και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Όπως σας είπα, ο βασικός ρόλος της νομικής υπηρεσίας στην Επιτροπή είναι το κριτήριο ε, του παραδεκτού, τα κριτήρια μάλλον για να γίνει μια παραδεκτή μια αναφορά, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε με νομική συνδρομή για να διαπιστώσουμε τι θα ήταν ε, και σωστό για συνέχεια μιας απόφασης. Η απόφαση που λαμβάνεται για μια αναφορά είναι πολιτική αναφορά ε, και υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών για να μπορέσετε να αποφασίσετε ε, τι προτιμάτε. Και εμείς φυσικά εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε στην παρακολούθηση, ιδίω αν αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Από διοικητική σκοπιάς η νομική υπηρεσία είναι μία από τις 13 γενικές διευθύνσεις ε, της ε, Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το βασικό καθήκον είναι να ε, δώσει συμβουλή στα, στους πολιτικές φορείς του Κοινοβουλίου. Τι προσπαθώ να πω. Η νομική υπηρεσία δεν δίνει συμβουλές στα μέλη, στους ευρωβουλευτές ξεχωριστά, αλλά στους πολιτικούς φορείς. Έχουμε μια ομάδα Είμαστε 75 νομικοί με εμπειρογνωμοσύνη σε όλη τη νομική παράδοση, και την ένομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε νομικούς από όλες τις εθνικότητες των κρατών μελών, οι οποίοι επιλέγονται και προσλαμβάνονται βάσει των ίδιων υψηλών απαιτήσεων ε, με τους υπόλοιπους ευρωϊπαλλήλους της Ένωσης με και το κριτήριο της ανεξαρτησίας και της επαγγελματικής ε, αρμοδιότητας φυσικά. Και κατόπιν ο τρόπος να λάβει κανείς συνδρομή από την νομική υπηρεσία συνοψίζεται στα εξής. Έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Ο παραδοσιακός τρόπος να διαβουλευτεί κανείς με την νομική υπηρεσία ε, είναι μέσω επίσημης γνώμης. Η επίσημη γνώμη μπορεί να ζητηθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής ή στην περίπτωση του Κοινοβουλίου και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Η διαβούλευση με την νομική υπηρεσία και οι κανόνες διαβούλευσης έχουν αποφασιστεί από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου στην απόφαση στις 28 Ιανουαρίου του 2004 που μπορεί η γραμματεία να στείλει σε όλα τα μέλη μετά από το τη της Αυτό το οποίο μπορείτε να δείτε σε αυτή την απόφαση είναι ότι οι ευρωβουλευτές μπορούν να ζητήσουν επίσημη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ε, αποστέλλοντας αίτημα ε, το οποίο θα απευθύνεται στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν όμως και ανεπίσημες συμβουλές ε, τις οποίες προσφέρουν οι νομικοί μας καθημερινά στι συνεδριάσει των επιτροπών, στι συνεδριάσει των συντονιστών, βοηθούν επίσης και τη γραμματεία να καταρτήσει το έργο της και ούτω καθεξής. Αλλά ως προς αυτό θα ήθελα να επισημανώ ότι η νομική υπηρεσία είναι υπηρεσία και εδώ ε, έχουμε την προστιθέμενη αξία μας ε, σε σχέση ε, με το συνδρομή ενός μόνο νομικού. Υπάρχει ο κίνδυνος βεβαίως κάποιες φορές, σπανίως, αλλά συμβαίνει και αυτό, οι συμβουλές οι οποίες προσφέρονται από τους νομικούς μας, σε αυτή την περίπτωση των εξαιρετικά καταρτισμένων τον κύριο Λικόνεν, να ε, έρχονται σε αντίθεση με την απόφαση της υπηρεσίας. Συμβαίνει σπανίως, αλλά είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε ευελιξία και ταυτόχρονα να έχουμε και την εμπειρογνωμοσύνη της ε, νομικής υπηρεσίας. Πρέπει επίσης να πω ότι δεν είμαστε τμήμα μελετών. Δεν έχουμε πόρους για κάτι τέτοιο. Ε, πολλοί από τους συναδέλφους πολλοί θα ήθελαν να κάνουν τέτοια δουλειά, αλλά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και επομένως η δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε με τα ε, νομικά προβλήματα για τις δυσκολίες που έχετε και όχι τεχνικά και ακαδημαϊκά ερωτήματα. Ζητώ ήδη την κατανόησή σας, ε, αν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Πολύ συχνά μας ζητούν ε, ε, πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε πόρους για κάτι τέτοιο. Δεν είναι θέμα διάθεσης, απλώς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα βασικά μας καθήκοντα. Και βεβαίως το μήνυμά μου σήμερα είναι απλό. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος να θέσει ερωτήσεις στην νομική υπηρεσία. Θα τα πω στα βουλγαρικά, λέει ο κύριος. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και το διοικητικό άχθος ε, είναι εθνική αρμοδιότητα. Αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο τη εθνική νομοθεσία. Όμω, οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, η ευρωπαϊκή νομοθεσία περιλαμβάνουν πολλέ κατευθυντήριε γραμμέ για την προώθηση των ε, μικρών οικογενειακών παραδοσιακών επιχειρήσεων. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Όταν η εθνική νομοθεσία ενό κράτου μέλου, ε, λέει ο κ. Κάνεν, στην προκειμένη περίπτωση για τη Βουλγαρία μιλώ, που έχουμε έναν κανονισμό που δεν αρέσει σε επιχειρήσεις γιατί κλείνει πολλούς μικρούς, ε, πολλά μικρά πρατήρια βενζίνης. Ε, όταν λοιπόν ε, πλήττονται ε, μικρές επιχειρήσεις προς όφελος μεγάλων υπάρχουν άλλοι τρόποι ώστε να υπάρξει προστασία για αυτές τις μικρές επιχειρήσεις από την Κομισιόν. Some member? Κάποιος άλλος? Ένα λεπτό να δώσω στην κυρία Μαρτίνεθ. Κοιτάξτε, είναι υποθετική η κατάσταση αυτή. Πάντως εντάσσεται ε, στα δικαιώματα και στη δραστηριότητα ουσιαστικά στη... στα όρια της, ε, και στα, δικαιώματα που έχει κάποιος για να υποβάλει μια αναφορά. Αν γίνει μια τέτοια αναφορά λοιπόν, θα κρυθεί παραδεκτή. Από εκεί πέρα θα δούμε τι μπορεί να γίνει βέβαια. And thank you to your... Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαρτίνεθ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και εσάς και την ομάδα σας ε, και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η παρουσίαση του θεματικού τμήματος Γ της συνεργασίας του με την Επιτροπή Αναφόρων. Ξέρετε ότι τα θεματικά τμήματα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις, κάτι που είναι αναγκαίο για τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μικέλ Τέλ που είναι ο προϊστάμενος της μονάδας θεματικού τμήματος ΓΑΜΑ για τη στήριξη και παροχή ειδικών συμβουλών για το τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ, αγαπητή Πρόεδρε. 5 λεπτά θα χρειαστώ για να σας παρουσιάσω το θεματικό τμήμα γάμα σαν τρεις γραμμές και έτσι να έχετε την ε, δυνατότητα, εφόσον θυμείτε, να θέσετε ερωτήσεις. Το θεματικό τμήμα, τα θεματικά τμήματα γενικά, είναι μια μονάδα μελέτης και έρευνας. Στηρίζουν το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τη χάραξη ομοθεσία, για την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την εκπλήρωση των γενικών ε, καθηκόντων και την, ανάθεση, την ανάληψη πρωτοβουλίων. Εμείς είμαστε ε, αρμόδιοι και για τα συνταγματικά θέματα και παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση και πληροφορίες σε επιτροπές με νομικό υπόβαθρο όπως είναι η ΛΥΜΠΕ, η Γιούρη, η ΑΦΚΟ, ΦΑΜ, Επιτροπή Αναφορών. Η μονάδα μας συνεργάζεται στενά με όλους ε, τους αρμοδίους ε, υπεύθυνους πολιτικής, ε, εισηγητές, γραμματεία από τις διάφορες επιτροπές, ώστε να έχουν επιτροπές ε, προσαρμοσμένες, ε, στοχευμένες, ποιοτικές, ανεξάρτητες, αμερόληπτες πληροφορίες ε, και ειδικέ γνώσεις, κάτι το οποίο θα στηρίξει τις ειδικές τους ανάγκες. Οι πολιτικοί αναλυτές που κάθονται εδώ δίπλα μου, σιγά σιγά θα τους γνωρίσετε, προσπαθούν να, να ενημερώνονται ε, ενημερώνονται για τη βιβλιογραφία από τις διάφορες πανεπιστημιακές πηγές, από τα διάφορα think tank κτλ. Άρα προσπαθούμε να ενημερωθούμε για την έρευνα που υπάρχει, για τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν και βλέπουμε πού ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη και σκόπιμη νέα έρευνα για την Επιτροπή σας και έπειτα βλέπουμε αν μπορούμε αυτό να το εξασφαλίσουμε εδώ εσωτερικά, δηλαδή μέσα στα δικά μας τα θεματικά τμήματα ή κάτι που είναι και σύνηθες, αν θα χρειαστεί να προσφύγουμε σε ξένους, ε, μάλλον σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Δεχεζόμαστε επίσης και τον προϋπολογισμό ε, για την έρευνα. Η δική σας επιτροπή έχει στη διάθεσή της 221.000 ευρώ. Το 2018 ήταν αυτό το ποσό διαθέσιμο, πολλά χρήματα σίγουρα, αλλά εμείς με αυτό το ποσό προσπαθήσαμε να κάνουμε και συγκριτικές μελέτες, κυρίως για να δούμε τι γίνεται σε 8-10 κράτη-μέλη. Και τέτοιου είδου μελέτε είναι δαπανηρέ συνήθω. Λοιπόν, διαχειριζόμαστε τον προπολογισμό αυτό με βάση τι κατευθυντήριε γραμμέ που αφορούν ε, την αμοιβόμενη εμπειρογνωμοσύνη. Είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ που έχουν εγκρίνει το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Ακολουθούμε και τη διαδικασία προκήρυξη διαγωνισμού όπω αυτή ορίζεται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Προσπαθούμε να επιλέξουμε πάντοτε του καλύτερου δυνατού εμπειρογνώμονε τη αγορά, εντό αγωγικών, αν μπορώ να μιλήσω για αγορά εδώ, φυσικά με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία. Και στόχος είναι να έχουμε και την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους ε, και προσφοράς, που δεν είναι πάντοτε εύκολο ή δεδομένο. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε στενά με αυτούς τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ε, τόσο ώστε η έρευνα που εσείς ζητείτε, που η Επιτροπή σας ζητεί, να ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες της. Προσπαθούμε στο έργο μας να είμαστε αμερόληπτοι, αντικειμενικοί και διαφανείς. Μαζί σας επίσης εκπονούμε την εντολή για τη μελέτη, ποιο είναι το πεδίο, ποιο είναι το περιεχόμενο. Πλησιώνουμε τους εμπειρογνώμενους στο έργο τους όλη τη διάρκεια αυτής της ε, μελέτης. Και έπειτα ερχόμαστε εδώ και σας παρουσιάζουμε τη μελέτη. Η έρευνα για κοινοβουλευτικούς σκοπούς έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έχει τις ιδιαιτερότητές της. Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα. Πρέπει να υπάρχει ακαδημαϊκή αριστεία, αυθεντία και να έχει ένα πρακτικό χαρακτήρα, να έχει δηλαδή μια χρησιμότητα η μελέτη, η έρευνα αυτή για την Επιτροπή σας και παράγουμε διάφορα προϊόντα ερευνητικού τύπου briefings, 10 σελίδες το πολύ, ε, σε βάθος αναλύσεις ε, από 11 36, 40 σελίδες και βέβαια μεγάλες μελέτες που υπερβαίνουν 40 σελίδες που στην προκειμένη περίπτωση είναι συγκριτικές μελέτες. Επίσης ε, σας προετοιμάζουμε και κάποια σεμινάρια για να εξετάσουν εκεί ζητήματα πολιτικής. Προσκαλούμε τους ε, καλύτερους κατά το δυνατόν εμπειρόνομες, τους ζητάμε να έχουν προετοιμάσει ένα σύντομο paper και έρχονται εδώ μετά και ε, συμμετέχουν σε μια ακρόαση. Επίσης, οι δημόσιες ακροάσεις ε, είναι ένα εργαλείο που έχετε εσείς στη διάθεσή σας. Βέβαια εκεί εσείς επιλέγετε τους εμπειρόνομους, ενώ στα εργαστήρια που βοηθούμε να διοργανωθούν επιλέγουμε εμείς τους καλύτερους κατ' εμάς εμπειρογνώμονες για να συζητήσω τα διάφορα θέματα. Πώς γίνεται λοιπόν ένα αίτημα, πώς κατατίθεται ένα αίτημα για έρευνα. Μόνο οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη. Εμείς είμαστε πιο ευέλικτη με την έρευνα που παράγουμε εμείς εσωτερικά εδώ στο Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη όταν εκπονούμε εκθέσεις ή κάποιο briefing για αποστολές ή αντιπροσωπείες. Και βέβαια αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το, όπως το αποκαλούμε, το ετήσιο ερευνητικό πρόγραμμα, Annual Research Program, που μόλις ε, άνοιξε, μόλις ξεκίνησε ε, να τρέχει προθεσμία για το πρόγραμμα αυτό, που είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε έγκαιρα έρευνα, εξωτερικέ μελέτες βέβαια, ιδίω όταν είναι μια μεγάλη μελέτη, παίρνει χρόνο. Δύο-τρει μήνε ή έξι μέχρι οκτώ μήνε. Γι' αυτό και αυτή η άσκηση για την εκπόνηση του ετήσιου ερευνητικού προγράμματος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς βλέπουμε το νομοθετικό πρόγραμμα της Προεδρίας, της Κομισιόν, τα, τα πολιτικά ψηφίσματα και ανάλογα προχωρούμε. Η Επιτροπή Αναφορών έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό βλέπουμε τον αριθμό αναφορών που έχουν παραληφθεί, τις γενικές αρμοδιότητες και το γενικό ενδιαφέρον, τα γενικά ενδιαφέροντα της Επιτροπής σας. Παραδείγματο χάρη, εκπονήσαμε μία μελέτη για το τι πέτυχε στην τελευταία θητεία η Επιτροπή Αναφορών. Θα δείτε ότι έχουμε μελέτες για τα δικαιώματα των παιδιών, πολλές μελέτες για το περιβάλλον, ενέργεια, με ρήπανση, διαχείριση υδάτων, επικίνδυνες ουσίες. Γιατί, διότι λάβαμε πάρα πολλές αναφορές επ' αυτών των θεμάτων και εσείς ζητήσατε πληροφορίες και εμπειρονομοσύνη για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τώρα έχει ε, ανοίξει η προθεσμία. Εμείς θα σας πλαισιώσουμε, θα συνεργαστούμε μαζί σε αυτή τη ε, διαδικασία και ελπίζουμε να έχουμε έτοιμο το ερευνητικό πρόγραμμα πριν τα τέλη Οκτωβρίου. Βέβαια, το ερευνητικό πρόγραμμα δεν ε, είναι κάτι που δεν μπορεί μετά να αλλάξει. Εσείς μπορείτε να ζητήσετε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ε, για επιπλέον ε, μελέτες, έρευνες και επίσης μπορούμε μέσα σε 5-6 μήνες να έχουμε αναθεωρήσει ίσως τροποποίησει το ερευνητικό πρόγραμμα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει όμως έστω στα τέλη Οκτωβρίου για να μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Αυτά είχα να σας πω. Αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε τον κύριο Τέιλ. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο. Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. σημείο που είναι η παρουσίαση της Έμιλι ε, Οράιλι της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την ετήσια έκθεση για το 2018. Κάθε χρόνο η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εκπονεί μια έκθεση για τις δραστηριότητες της η οποία παρουσιάζεται επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που υποβάλλεται και στην Επιτροπή Αναφορών. Η ετήσια έκθεση του 2018 δημοσιεύθηκε μεν το Μάιο, αλλά υποβάλλεται στην Επιτροπή Αναφορών ε, λόγω της διακοπής ε, των ε, δραστηριοτήτων και των ευρωεκλογών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κάθε χρόνο, θα εκπονήσει έκθεση για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και τις δραστηριότητες του 2018. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Πίτερ Γιάρ από το ΕΛΚ, ο οποίος θα υποβάλει την έκθεσή του στη συνεδρία του Οκτωβρίου. And we are going to wait. Περιμένουμε τώρα λίγο. The ombudsman. But we are going to go on time. I'm sure. Αλλά θα προλάβουμε και θα γίνουν όλα γέρος. Είμαι βέβαιη. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Ωραϊλή. σας περιμέναμε. Πρέπει να τελειώσουμε στις 12 με το δικό σας θέμα. Αν, αν συμφωνείτε θα σας δώσω 10 λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για, τις, ε, για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι στην Επιτροπή και γνωρίζω και τα μέλη ε, τα καινούρια. Ε, θα σας παρουσιάσω λοιπόν την έκθεσή μου για το 2019, του 2019, κοιτώντας το 2018 να δούμε τις βασικές υποθέσεις, πώς συνεργαστήκαμε με αυτή την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα. Σύντομα, κάποιοι από εσά μπορεί να μην γνωρίζετε την, ε, τον θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που εκλέγεται από το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν έχουν να κάνουν με αυτό. Δεν σε ε, θέτει ως υποψήφιο η χώρα σου. Ε, είσαι άτομο ξεχωριστό, ανεξάρτητο και θέτεις υποψηφιότητα βάσει της δικής σου καριέρας. Ε, αντιμετωπίζω προσφυγές ε, για θέματα που έχουν να κάνουν με τα θεσμικά όργανα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, δεν έχω να κάνω με, με δεν έχουμε αντικ, αντικρώμενα ας πούμε, συμφέροντα γιατί εσείς ασχολείστε με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Εγώ κάνω συστάσεις, δεν είμαι δικαστής που αποφασίζει, όμως το 85 περίπου των συστάσεών μας ε, έγιναν δεκτές. Αυτό είναι καλό, θεωρώ. Επίσης, οι εξουσίες. Μπορώ να εξετάσω οποιοδήποτε έγγραφο ε, θέλω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσω ότι ξέρω όλα τα γεγονότα σε σχέση με μια αναφορά ε, μπορώ να δω οποιοδήποτε έγγραφο, όσο εμπιστευτικό και αν είναι, φυσικά δεν μπορώ να το δημοσιεύσω. Επίσης μπορώ να καλέσω ως μάρτυρες ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μπορεί και από μόνη μου, με δική μου πρωτοβουλία, να κάνω μια έρευνα Υποπτεύομαι ότι υπάρχει ένα θέμα που θα έπρεπε να διερευνήσω ακόμα και αν δεν είχα συγκεκριμένο παράπονο, συγκεκριμένη προσφυγή γι' αυτό. συνεργάζομαι με το Κοινοβούλιο πολύ στενά, ειδικά με αυτή την Επιτροπή, στην οποία λογοδοτώ κυρίω. Θα δείτε επίσης και άλλες επιτροπές τι οποίε πήγα το 2018 φυσικά και στην Ολομέλεια αλλά και στη διάσκεψη των Προέδρων και των Προέδρων των Επιτροπών. Επίσης ε, είχα συναλλαγές ε, και συνομιλίες ε, λόγω των προσφυγών από ευρωβουλευτές που είναι πολύ χρήσιμες ε, γιατί βελτιώνεται η διοίκηση. Υπάρχει πάντοτε ένα στοιχείο δημοσίου συμφέροντος σε αυτές. Γι' αυτό ε, γενικά το 2018 αντιμετωπίσαμε 2.180 προσφυγές. Είχαμε αύξηση κατά 17% των προσφυγών που ήταν εντός της εντολής μας, 880 συνολικά. Είναι καλό αυτό γιατί πλέον υπάρχει μια εμπειρία. Αυτές που είναι εκτός εντολής είναι συνήθως αυτές με τις οποίες ασχολείται ε, ο κρατικός, ε, ο διαμεσολαβητής, ο συνήγορος του πολίτη σε κάθε κράτος μέλος ή η επιτροπή σας ε, για να μπορέσει ο πολίτης να βρει μια λύση για το πρόβλημά του. Ε, είναι οι περιπτώσεις, η διαφάνεια, πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έγγραφα, αυτά είναι σημαντικά θέματα για μας, τα θεμελιώδη δικαιώματα, αν υπάρχουν ας πούμε αιτιάσεις ότι δεν γίνονται σεβαστά, συμμετοχή των πολιτών σε δημόσιες διαβουλεύσεις, σε ε, πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών, τέτοια θέματα. Επίσης, προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. πολλές φορές έχουμε παράπονα ότι η Κομισιόν έχει δώσει χρήματα σε ένα άτομο ή μια ομάδα και τα χρήματα που δόθηκαν δεν δαπανήθηκαν σωστά, π.χ. έρχονται σε εμά και κοιτάμε ακριβώς ποια είναι η ιστορία, ποιο είναι το ιστορικό και αν υπάρχει κάποια επίσης σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για μας, ε, όσον αφορά δηλαδή επιτρόπους, ε, μέλη του προσωπικού, ε, συμβούλους, εμπειρογνώμονες. Κοιτάζουμε λίγο αυτά τα στοιχεία, αλλά και κάποια θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, π.χ. καθυστερήσεις και περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχε σωστή μεταχείριση κτλ. Από πού παίρνουμε τις περισσότερες αναφορές. Για πού μάλλον. Ε, κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή είναι το πιο δραστήριο όργανο, όχι επειδή είναι κακή η διοίκηση, απλώς έχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με το κοινό. Και μετά έχουμε το κοινοβούλιο, όχι ως προς τον πολιτικό του ρόλο, αλλά ως προς τον διοικητικό του ρόλο. Μετά έχουμε, και τα βλέπετε και στο PowerPoint που σας δώσαμε, παραδείγματα για τα ε, για τις επιληθήσεις ε, προσφυγές το 2018, ας πούμε, μια χορήγηση που δόθηκε σε μια ερευνητική εταιρεία από την Κροατία ε, για παράκτιες έρευνες. Η Κομισιόν προσπάθησε να πάρει πίσω 700.000 ευρώ. Όταν όμως εξετάσαμε εμείς το θέμα, το ποσό μειώθηκε στα 300.000 ευρώ. Το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων έχει να κάνει συνήθως ε, με το πώς ελέγχονται τα φάρμακα, την πρόσβαση στα έγγραφα. Εδώ είχαμε μια υπόθεση σε σχέση με μια εταιρεία που είχε ζητήσει πρόσβαση σε μια έκθεση ε, ασφαλείας, ενημέρωση ασφαλείας για ένα φάρμακο. Και εδώ θα δείτε και κάποια άλλα παραδείγματα. Ένα Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων, άλλο ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Η Κομισιόν τους πλήρωσε τα χρήματα που ήταν υπό αμφισβήτηση. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε επίσης και ζητήματα όπως ε, τον διορισμό του πρώην Γενικού ε, Γραμματέα την Επιτροπή, ε, τα γνωρίζετε ακόμα και εσείς που δεν είστε καινούργοι, είναι θέματα που ερευνούμε, ερευνούμε το, όχι το άτομο όμως, αλλά το πώς η Κομισιόν αντιμετωπίζει το θέμα. Είχαμε τέσσερις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και η σύσταση ήταν να υπάρχει διαφορετική διαδικασία για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή βέβαια απέρριψε τη σύστασή μας, αλλά θα υπάρχει νέα Επιτροπή, νέος Γενικός Γραμματέας σύντομα και θα δούμε ακριβώς πώς θα διενεργηθεί η διαδικασία σε αυτή την περίπτωση και θα έχουμε δεχομένως τελικά μια θετική αντίδραση στην σύστασή μας. Στρατηγική εργασία το 2018 πώς κάνουμε αυτές τις έρευνες. Χρειαζόμαστε πολλές πληροφορίες. Δεν είμαστε τόσο πολύ εκεί για να επικρίνουμε, αλλά για να βοηθήσουμε εμείς στην Κομισιόν και στα άλλα θεσμικά όργανα ή γραφεία ή οργανισμούς, παρουσιάζουμε τον τρόπο που μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα για να μην λαμβάνουν προσφυγές. Γιατί πολλές φορές δεν το έχουν σκεφτεί και πολλές φορές μας ευχαριστούν για τη δουλειά που κάναμε, για το πώς επιλύσαμε το πρόβλημά τους. Να, κάποια στρατηγική δουλειά που κάνουμε το 2018. Η πρόκληση της αυτόματης πόρτας για, τις για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Φαίνεται ότι κάποιοι τομείς ε, φεύγουν από το δημόσιο τομέα και πάνε στον ιδιωτικό. Απλώς ε, δεν πρέπει να φύγετε το δημόσιο συμφέρον. Αυτό εμείς προσπαθούμε να φροντίσουμε επίσης ε, προς παρασκευαστικές διαδικασίες ε, για εγκρίσεις φαρμάκων, ε, κάποια προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, μηχανισμοί προσφυγών για τα διαρθρωτικά ταμεία και για το Brexit η διαδικασία του άρθρου 50. Προσπαθήσαμε να δούμε ότι υπήρχε διαφάνεια σε αυτό. Κάτι άλλο τα τελευταία χρόνια που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η λογοδοσία του Συμβουλίου. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθούν τις νομοθεσίες, μπορούν να παρεμβαίνουν, προσπαθούν να τις επηρεάσουν. Εμείς αυτό που εξετάσαμε ήταν πόσο διαφανές ήταν το Συμβούλιο σε σχέση με την νομοθετική διαδικασία. Κάναμε, ας πούμε, μια έτσι, αστυνομική δουλειά. Ψάξαμε έγγραφα, είδαμε πώς λειτουργεί η διαδικασία και βρήκαμε κακοδιαχείριση, έλλειψη δηλαδή διαφάνειας και κάναμε συστάσεις για το πώς μπορεί αυτό να απαλληλθεί καταγραφή των θέσεων π.χ. των κρατών μελών, καθώς προχωρά η νομοθεσία, δεν λέμε να δημοσιεύονται, αλλά να καταγράφονται σίγουρα. Και για να διασφαλίσουμε ε, ότι ε, δεν γίνονται αυτόματα εμπιστευτικά όλα τα έγγραφα που βγαίνουν. Κάποια μπορεί να ε, είναι πιο ελεύθερα, αν είμαστε από πριν εκεί και προλαμβάνουμε τις διαδικασίες. Βέβαια, το Συμβούλιο δεν είχε την απάντηση που θέλαμε και την αντίδραση που επιθυμούσαμε για αυτό το θέμα. Κάναμε λοιπόν μια ειδική έκθεση πέρυσι στο Κοινοβούλιο και είχαμε την ε, υποστήριξη μεγάλη, της μεγάλης πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλοί που μας υποστηρίζουν σε αυτό. Αργότερα, μέσα στο, μέσα στο μήνα, θα συναντηθώ με τον Δανό Πρωθυπουργό, αλλά και η Φινλανδική Προεδρία θα προωθήσει το θέμα. Ένα κομμάτι ας πούμε, της λογικής που χρησιμοποίησαμε σε αυτή την έκθεση ήταν να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα που ε, έχει το γεγονός ότι οι πολίτες ε, δεν κατανοούν πόση επιρροή έχουν τα κράτη τους ε, στην νομοθεσία που βγαίνει από τις Βρυξέλλες και κατηγορούν συνέχεια τις Βρυξέλλες. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας το 2018 ήταν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Συνηγόρων του Πολίτη, των Διαμεσολαβητών. Ήρθαν όλοι στις Βρυξέλλες ε, για σεμινάριο και μπορέσαμε να συνομιλήσουν με διάφορους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανώτατα στελέχη και είδαμε πώς θα υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους, ε, ποιος ε, θα βοηθάει ποιον, αν υπάρχει δυνατότητα εμείς να βοηθάμε τις περιφερειακές υπηρεσίες ε, και πώς θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Και τέλος, το ευχάριστο κομμάτι της δουλειάς μου. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύουμε για την καλή διοίκηση, Μπορώ να πω ότι μπορούμε πια να χαιρόμαστε για το ότι υπάρχουν καλές πρακτικές, μπορούμε να τις μοιραστούμε. Πριν από μερικές μέρες δώσαμε κάποια βραβεία, ας πούμε, ε, καλής διοίκησης ε, και αυτό ήταν ένας ωραίος τρόπος να δώσουμε ένα ευτυχισμένο τέλος σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Οράιλη για τις εκτεταμένες εξηγήσεις που δώσατε για την έκθεση που μας παρουσιάσατε. Θέλει κάποιος να μιλήσει, παρακαλώ, η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για τη δουλειά σας η οποία είναι αξιοθαύμαστη πραγματικά. Πόσα κάνετε και τα αποτελέσματα. Ορισμένες φορές ε, ε, απογοητεύομαι, ε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εσείς δίνετε τη μάχη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσετε κάποια θέματα. Δύο πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχει ακόμα επιληθεί το θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν από το κόμμα μου, αλλά ξέρετε, ορισμένες φορές ε, το συγχέουν με τα συμφέροντα και τις εξουσίες των ευρωβουλευτών. Το, η σύγκρουση συμφερόντων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ε, να ε, εξετάσουμε, διότι αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις ε, ε βάσει νόμου για το, η ζωή των πολιτών. Είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τουλάχιστον στη χώρα μου, και αυτό ισχύει σε πολλές χώρες. Δεν έχει ακόμα κανείς αντιληφθεί τι ακριβώς είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά, πιστεύω, επί του θέματος, για να μπορέσουμε να έχουμε και σωστή διαχείριση. Και μετά, για τη διαφάνεια του Συμβουλίου, όπου βεβαίως ε, καλωσορίζουμε πάρα πολύ τα όσα έγιναν. Υπήρχε και μια αναφορά από τους πρασίνους ε, για την κοινή απάντηση που λάβαμε με την ΑΦΚΟ στην εκθεσή ε, σας, η κυρία Τόμ, ε, ο Γιώ Λάινεν και λάβατε πλήρη υποστήριξη. Και εδώ ανησυχώ λίγο. Διότι αν δω τις, αποφάσεις, τις απαντήσεις των κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής μου, της δανέσκης κυβέρνησης, ε, πάντα όλοι λένε «Α, χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω διαφάνεια», χωρίς να αντιλαμβάνονται βασικά αυτό που λέει η έκθεσή σας, που λέει ότι φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι διακυβερνητικός οργανισμός ε, είναι διεθνή οργανισμό. Ε, όλοι είναι διεθνείς οργανισμοί, έχουν διπλωμάτες και εργάζονται έτσι. Φέτος, είναι ένα οργανισμό που νομαθετεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν δικαίωμα τα εθνικά κοινοβούλια και ο εθνικό τύπο να μπορούν να παρακολουθήσουν τι κάνει η κυβέρνησή τους και σε όλες τις επιτροπές. Και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και λέω εμείς γιατί είναι κοινή η πρόκληση. Ε, θέματα εξωτερικής πολιτικής ε, ε, βρίσκονται σε πολύ δυσάρεστη θέση με κάτι τέτοιο. Ο κόσμος πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τι γίνεται. Εμείς είμαστε, αυτοί είναι συνηθισμένοι να δουλεύουν μυστικά, χωρίς να μαθαίνουν τα πράγματα παρά έξω. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, να μην καλωσορίζουμε κάποια καλά ωραία λόγια για το να έχουμε περισσότερα έγγραφα και λιγότερα γραφειοκρατία και να μην βάζουμε τη σφραγίδα της εμπιστευτικότητας παντού, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι στην ημερήσια διάταξη και μετά στα πρακτικά και πώς ε, ε, ε τοποθετήθηκε η τάδε ή δύνατη προσωπία ε, για να μπορέσετε κι εσείς να το δείτε και στην έκθεσή σας για, όπως το λέτε να υπάρχει λογοδοσία για ό,τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά αυτό ισχύει για το Συμβούλιο. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί νομίζω ότι ακόμα πάσχουμε από κάτι που δεν το αντιλαμβάνεται ούτε καν ο κόσμο στο κοινοβούλιο. Θεωρούν ότι δεν πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Υπάρχει δηλαδή κάπου ένα κενό, ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Ε, και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε σωστά το έργο του Συμβουλίου. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω πρέπει να είμαστε πιο σκληροί. Και αν το Συμβούλιο συνεχίσει να αρνείται ε, να, ε, ε, διορθώσει αυτό το θέμα, υπάρχει δυνατότητα να προσφύγουμε στο δικαστήριο εναντίον του. Εσεί, πολύ σωστά, δεν αναφέρεστε στο 1049 στην νομοθεσία, αναφέρεστε στη συνθήκη και λέτε ότι αυτό είναι παραβίαση των βασικών αρχών τη συνθήκη. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Είναι σοβαρό δεν είναι το πώς ερμηνεύουμε το 1049 και τι εξαιρέσει πρέπει να έχει κλπ. Είναι πιο ουσιαστικό. Ίσως είναι πολύ δύσκολο για σας ε, να μας πείτε και τι θα πρέπει να κάνουμε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να καθόμαστε εδώ άπραγοι και να εγκρίνουμε και να συμφωνούμε με αυτό που λέτε «Α, είναι παραβίαση της και μετά να μην κάνουμε τίποτα. Κάπως πρέπει να το συνεχίσουμε. Κυρία Όκεν, έχει και άλλα μέλη που θέλουν να λάβουν το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Πίτερ Γιάρ. Ah, Πάλι με το μικρόφωνο έχω πρόβλημα. Έξι είχα σημειώσει στο χαρτί μου. Να πω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και γι' αυτό και για την καλή συνεργασία με την Επιτροπή ε, Αναφορών ε, που ήταν πολύ επικοδομητική. Το δεύτερο είναι αν χρειαζόμαστε Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Νομίζω ότι ναι, το έδειξε και η ε, παρεμβασή σα με τι καταγγελίε που λαμβάνετε. Πολλοί στρέφονται σε εσά, Αυτό είναι σημαντικό και έτσι πρέπει να ισχύει σε μια δημοκρατία. και σίγουρα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ε, ε, του τι γίνεται σε μια δημοκρατία. Είπατε ότι δεν υπάρχει επαρκέ διαφάνεια στο Συμβούλιο και τι κάνετε επ' αυτού. Και εμεί πρέπει ε, επ' αυτού να αντιδράσουμε γιατί υπάρχει αδιαφάνεια και στη Γερμανία σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Εκεί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα και παρόλα αυτά είχε ψηφίσει η Γερμανία στο Συμβούλιο, τα πίεσε, αλλά δεν εφαρμόζονται και γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και είναι καλό το ότι ε, τα συζητούμε και ότι δεν είναι σε εύκολη θέση το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή λόγω αυτών των συζητήσεων. Αυτό είναι θετικό και είναι ένα θετικό παράδειγμα. Το Κοινοβούλιο έχουμε διαφάνεια ε, υπάρχουν σίγουρα κάποια σημεία που δεν είναι τόσο ε, δημόσια, αλλά νομίζω ότι το Συμβούλιο είναι ένα κακό παράδειγμα. Και το τελευταίο σημείο, κύριε Ράιλι, Θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία και σας και στον υποψήφιο για την επόμενη θητεία, γιατί η εκλογές είναι το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Έμιλι για την ε, εργασία σας και για την παρέμβασή. Συμφωνώ και εγώ με τον Πίτερ ότι φαίνεται από την παρέμβασή σας σήμερα και από το έργο που έχετε κάνει πόσο σημαντική είναι η αρχή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ε, όχι για να έχουμε ε, απλά μια αυτοκριτική στο πώς δουλεύουν τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά γενικότερα το πρώτο σημείο που θέλω να σχολιάσω αναπόφευκτα είναι το Brexit. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ θετικό και από τη Βρετανική κοινή γνώμη το ότι υπήρξε τόσο μεγάλη διαφάνεια από τους ε, Ευρωπαίους διαμεσολαβητές, ε, κάτι που έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με το τι έκαναν οι Βρετανοί διαμεσολαβητές, ε, που δεν ε, ενημέρωναν καθόλου την κοινή γνώμη. Δηλαδή η Βρετανική κυβέρνηση ήταν πλήρως αδιαφανής ό,τι αφορά τη στρατηγική και για την προετοιμασία σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Αν συγκρίνουμε την διαφάνεια που υπήρξε από ευρωπαϊκή πλευρά για το τι προβλέπεται, ποια ήταν αλλακτικά σχέδια, αν υπάρξει no deal κτλ. Όλα αυτά ήταν ε, στη δημόσια ήταν δημόσια γνωστά στην κοινή γνώμη από τον Μισελ Μπαρνιέ και την πρακτευτική του ομάδα που πρέπει να το συγχαρούμε. Να το παραβάλουμε αυτό με εντελώς ε, ετερόκλητους ε, ετερόκλητες ανακοινώσεις 170 ε, διαφορετικές ροές εργασίας ε, στο, ε, από την πλευρά της Βρετανίας και καμία διαφάνεια για το τι συζητεί και προβλέπεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια στο Συμβούλιο, το ζούμε. Ζούμε το αποτέλεσμα δεκαετιών παραπληροφόρησης και ψευδών ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκεί, στην παραπληροφόρηση δηλαδή και στα ψεύδη, βασίστηκε ε, και η εκστρατεία του δημοψηφίσματος για το Brexit. Ε, 95% των αποφάσεων του Συμβουλίου. Το Ηνωμένο Βασιλείο συντασσόταν με την πλειοψηφία, δεν καταψήφιζε. Οι Βρετανοί υπουργοί έχουν συνυπογράψει πάρα πολλά νομοθετήματα. Επομένω, η διαφάνεια στο Συμβούλιο για μένα είναι κάτι θεμελιώδε για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματο και για την αξιοπιστία. Και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει την πραξιακή απειλή το Συμβούλιο από την αδράνεια το χαρακτηρίζει. Αυτό που είπε η Μάγκριτα το σημειώνω. Ίσως η μελλοντική συζήτηση θα έπρεπε να έχει ως θέμα τι θα γίνει ε, από εμά αν δεν αντιδράσει το Συμβούλιο. Τώρα, το δίκτυο των ε, συνηγορών του πολιτή είναι ένα ε, μέσο, ένα εργαλείο για να μπορεί να ασκεί βάση πίεση ώστε περισσότερες κυβερνήσεις στο Συμβούλιο να γίνουν περισσότερο διαφανείς μας παρουσιάσατε ε, το δίκτυο αυτών των συνηγόρων του πολίτη, αλλά δεν ακούσαμε κάποιες συστάσεις. Τι συζητείτε ε, σε αυτό το δίκτυο. Θα ήταν ενδιαφέρον. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα στη Διαμεσολαμήτρια. Να συγχαρώ και εγώ ε, την διαμεσολαβήτρια για την έκθεσή τη, όπω πάντα μα δίνει μια σαφή εικόνα των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε ώστε να υπηρετήσουμε με το σωστότερο δυνατό τρόπο τους Ευρωπαίους πολίτες. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δουλειά σας, ιδιαίτερα στην προάσπιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό που διαπίστωσα αναλύοντας τις τρεις ε, εκθέσεις των προηγούμενων ετών, κάνοντας δηλαδή μια συγκριτική ανάλυση, ε, είναι δυστυχώ μια πολύ αρνητική τάση και επονίδιστο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση και την ε, ε ε, αποστολή των συστάσεων έχει μειωθεί πάρα πολύ στην τελευταία τριωτία. Το 2018 το αναφέρατε κι εσείς, αλλά εγώ θα ήθελα να το ξαναπώ. Υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις ε, οι οποίες ε, σας απασχόλησαν και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπήρξε καμία απάντηση ή μάλλον δεν υπήρξε σαφής απάντηση. Ε, σε συνέχεια, για παράδειγμα, ε, από του σκανδάλου Σελμάιερ, του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, του Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγγνώμη, Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια για να υπάρξει μια νέα διαδικασία διορισμού και έτσι παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας, δεοντολογίας και κράτους δικαίου. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ μεγάλα κενά δεοντολογίας στι σχέσεις με τα ιδιωτικά λόμπι και το γεγονό ότι πολλοί φεύγουν και πηγαίνουν από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα ε, χωρίς να υπάρχει σύγκρουση, να θεωρείται ότι υπάρχει σύγκρουση συμφωνών. Και επίση αρνούνται να δώσουν πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτε, παραβιάζοντα τι βασικέ αρχέ τη διαφάνεια και τη διαφήμιση. Εγώ ελπίζω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αυτή τη νέα μάλλον Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία, η οποία θα βασίζεται στην εφαρμογή των υψηλότερων δεοντολογικών και ηθικών προτύπων και διαφα... της υψηλότερης διαφάνειας. Και θεωρώ ε, ότι ε, θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε ε, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας βοηθήσει ώστε να είναι όλο ένα και πιο δυσμευτικές οι συμβάσεις σας, οι, συ, οι συγγνώμη, και ε, να είναι και πιο εύρωστες. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο δουλέψατε, η διαφάνεια για το Συμβούλιο και εμείς πρέπει να μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα και να δώσουμε απαντήσεις στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ποιος μπορεί να είναι λοιπόν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να βοηθήσει έτσι ε, περισσότερο σε αυτά που έχετε να πείτε. Η κυρία Μπεντρέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Διαμεσολαβήτρα, Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας και τη δουλειά που έχετε διεξάγει ο ρόλος σας ήταν πολύ σημαντικός ε, για να αντιμετωπίσουμε το ρόλο του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για το δεσμό μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων και των πολιτών. 85% των συστάσεων είπατε ότι έχουν εφαρμοστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για τα συμβούλια και συγκεκριμένα για το ποιο ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που καταφέρατε το τελευταίο διάστημα και ποιο θέμα αντιθέτως, ποιο ήταν το πρόβλημα που είχατε κυρίως. Και πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένη δική μας Επιτροπή μπορεί να σας υποστηρίξει στη δουλειά σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ε, δίνω τα 30 δευτερόλεπτα. Όχι, δύο λεπτά. Ε, ε πρέπει να τελειώσουμε στις 12. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις, τα σχόλια. Θα τα απαντήσω σύντομα. Κυρία Άουκεν, όντως ε, συνεχίζεται αυτό το θέμα της σύγκρουση ε, συμφερόντων. Είναι θέμα κουλτούρας, θα έλεγα. Ε, σιγά σιγά αλλάζει. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα χρειάζεται ένα συνασπισμός ε, δυνάμεων για να αλλάξει το κοινοβούλιο και εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα πρέπει και η Επιτροπή να κάνει τη δική της ε, δουλειά. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε πρόοδο. Τώρα όσον αφορά στον κύριο Γιάρ και κυρία Άουκεν ε, για την νομιμότητα του Συμβουλίου και η κυρία Ντάρινγκ το ανέφερε. Συναντήθηκα με τον Φινλανδό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων χθε για να δω ποια είναι η πρόοδο στο Συμβούλιο και ποια είναι τα σχέδια που έχει η Προεδρία τους και αναγνώρισε τις προκλήσεις. Ρωτούν όμως και ζητούν από μένα να τους πω ποια είναι τα καλύτερα επιχειρήματα που μπορούμε να του δώσουμε. Είπατε κι εσείς για το Brexit, η έλλειψη γνώσης και ευαισθητοποίησης του ε, ε, κοινού στην Βρετανία άφησε αυτό το κενό ε, που έδωσε χώρο για να υπάρξει παραπληροφόρηση. Αυτά είναι τα θέματα της νομιμότητας ε, και αυτά είναι και τα ε, επιχειρήματα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εμπλέκονται στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κάνουν και στα κράτη-μέλη, στο χώρα τους δηλαδή. για το ευρωπαϊκά δίκτυα ε, συνηγόρων του πολίτη και το Brexit ε, να πω ότι έχω έρθει σε επαφή με τους ε, συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που ζουν σε αυτές τις χώρες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει πάντοτε αυτή η συζήτηση του τι θα γίνει όταν συμβεί το Brexit. Είπαμε ότι θα συνεργαστούμε για να δούμε τι θα γίνει με τους πολίτες που θα μείνουν ξεκρέμαστοι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δίκτυο για να προωθήσουμε τη διαφάνεια στο Συμβούλιο, βέβαια, είναι μια εξαιρετική ιδέα και σας ευχαριστώ για αυτό, κυρία Εύη. Ε, ευχαριστώ και πάλι ε, ως προς την περίπτωση του κυρίου Σαλμαϊέρ, του Γενικού Γραμματέα. Είπατε ότι δεν την παρακολουθήσαμε. Την παρακολουθήσαμε, απλώς είπαν όχι. Μας αγνόησαν. Το βασικό θέμα εκεί και το πρόβλημα ήτανε ότι φύγαμε από τον ουδέτερο χώρο της διοίκησης και πήγαμε σε ένα πιο σε πολιτικό επίπεδο, σε μια πολιτική σφαίρα. Αυτή ήταν η δυσκολία. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη. Με την νέα επιτροπή, με το νέο γενικό γραμματέα που θα διοριστεί, είμαι σίγουρη και από αυτά που είπε και η κυρία Φοντερ Λάιεν στην δική της ε, ομιλία, ε, όταν διορίστηκε ο Σινέα πρόεδρος της Επιτροπής, ε, είμαι σίγουρη ότι αυτά τα θέματα της διαφάνειας ε, θα έρθουν, ότι θα δούμε μάλλον αλλαγή. Τώρα, σε σχέση με το τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε πριν από χρόνια, γενικά ήμασταν επιτυχημένοι σε αυτά που κάναμε. Έχουμε πιο διαφανείς και διαδικασίες, υπάρχει περισσότερη ορατότητα ε, και πολλές από τις ε, προσφυγές είχαν σημαντικό ε, μια σημαντική διάσταση δημοσίου συμφέροντος για την ευρύτερη κοινωνία και αυτό είναι καλό. Είχαμε το κίνημα των συζύγων, ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ συνεχώς με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και είχαμε και εξαιρετική συνεργασία με αυτή την Επιτροπή, όπως και με άλλες. Οπότε με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Thank Σας ευχαριστώ όλους. Thank you very Pasamos al punto 9. Περνάμε στο σημείο 9. Que es la primera petición del día, que es la... Που είναι η πρώτη αναφορά της ημέρας. Πρόκειται για την 0596 του 2018 ε, του Μάρα Ισπανικής Ιθακένωσης εξ ονόματος της ε, ΑΕΠΣΙΣΙΕ σχετικά με τον καθορισμό μια ενωσιακή στρατηγική για τα διασταμικά καιρικά φαινόμενα και του ηλεκτρομαγνητικού παλμού. Να δώσουμε το λόγο στον αναφέροντα για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ και καλώ ορίσατε. Καλημέρα σα. Ως οργάνωση πολιτική Προστασία θέλουμε η παρέμβασή μα να απευθύνεται στου ανθρώπου που αντιμετωπίζουν τον όριο. Μισό λεπτό περιμένετε. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, να αποχωρήσουν ησύχω για να ακούσουμε και τον αναφέροντα. Ευχαριστώ. Έλεγα καλημέρα και ως οργάνωση πολιτικής προστασίας τα πρώτα λόγια ε, απευθύνονται σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πλήττονται ε, από τον Όριαν, ε, τους πληγέντες και τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας που δρούν αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Να Αναφερθούμε επίσης στους ε, μα, τον Χωσέ Σαβούρε Καμπέλ, ο οποίο ε, ε, προώθησε αυτή την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρώσουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε μόνο πέντε λεπτά και το θέμα της απειλής των ηλεκτρονικών παλμών είναι πολύ ευρύ και πολύ περίπλοκο. Γι' αυτό ζητούμε να εκπονηθεί μια στρατηγική τη Ένωση, στου δύο έξονες για τα καιρικά φαινόμενα και επίσης τα τεχνητά φαινόμενα, δηλαδή ω όπλο μαζικής καταστροφής. Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και να διευκρινίσουμε κάποιες έννοιες αν το θεωρεί η κατάλληλη Προεδρία. Κατά τα άλλα σας παραπέμπουμε στην ε, ε, τεκμηρίωση που σας έχουμε στείλει και εδώ θα αναφέρουμε πέντε σημεία πολύ συγκεκριμένα. το ηλεκτρονικό παλμός είναι ε, ταχύτατη εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που είναι ικανή να καταστρέψει τα πάντα. Ε, ο οργανισμός μας δεν αμφισβητεί την ευρωπαϊκή έρευνα σε θέματα φυσικών καιρικών φαινόμενων ή διαστομικών φαινομένων και αυτό το τονίζουμε. Είπαμε σαφώς ότι αυτό που λείπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άλλα πράγματα. Δεν είναι οι έρευνε αλλά σχέδια πολιτικής προστασίας και συντονισμού για αυτό το εξαιρετικό σενάριο το οποίο όμως μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο τη ηλεκτρομαγνητικής ακτιβολίας αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα ακραίο ηλιακό φαινόμενο, πολύ φυσικό, και αν ξεκινήσει έχουμε ελάχιστε ώρε μέχρι την, ε, τον αντίκτυπο και αν είναι διαστημικό έχουμε κάποια λεπτά. Αν τα σχέδια πολιτική προστασία δεν έχουν εκπονηθεί πριν από την έναρξη ενό τέτοιου φαινομένου, αυτή τη στιγμή ξεκινήσει με ελάχιστε ώρε περιθώριου ελιγμών, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι είναι τα πράγματα. Η επιστημονική έρευνα που υπάρχει είναι. Ε, ε, αξιοσημειωτή, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει αν δεν υπάρχει πολιτική προστασία και σχέδια πολιτική προστασία, τα οποία δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Ζητούμε λοιπόν μια πολιτική για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Δεύτερον, στην αναφορά μα είπαμε ότι στην Ευρώπη είμαστε 10 χρόνια πίσω στη ε, θέματα αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου και ε, η πρώτη επιτροπή EMP δημιουργήθηκε από τι Ηνωμένες Πολιτείε το 2001 και το 2009 συστήθηκε η πρώτη ε, επιτροπή από το Κοινοβούλιο των Ηνωμένων των ε, ΗΠΑ και αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν 20 χρόνια καθυστέρηση για την πρόληψη του συγκεκριμένου κινδύνου. Και αυτά δεν είναι απλά λόγια. Θα σα δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για να έχετε μια εικόνα του τι ακριβώ ε, συμβαίνει και το γεγονό ότι δεν έχουμε τίποτα. Η Επιτροπή Ρύθμιση Ενέργεια ε, το 2013 εξέδωσε το διάταγμα 779 που ζήτησε από όλου του ηλεκτρικού παρόχου τα πρότυπα ανάκτηση σε περίπτωση ενό ακραίου ηλεκτρομαγνητικού φαινομένου, είτε φυσικού είτε τεχνητού. Ε, μετά υπήρχε και δεύτερο διάταγμα σε δύο χρόνια, το 830. Δύο διατάγματα τα οποία αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το θέμα? Καμία. Οι δικοί μας υπάροχοι τι πρέπει να κάνουν σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση ενός παγκόσμιου τέτοιου φυσικού φαινομένου, να αυτοσχεδιάσουν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προχώρησαν. Ολοκληρώθηκαν και τα δύο το 2015. Ε, πριν από τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκε ο καθορισμό τη Εθνική Στρατηγική για τα διαστημικά θέματα και εμεί τώρα ζητάμε να αρχίσουμε να την καθορίζουμε τη στρατηγική. Πού είναι η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Οκτώβριο του 2016 υπήρχε ένα προεδρικό διάστημα από τον πρόεδρο Ομπάμα και το 2019 είχαμε άλλο προεδρικό διάταγμα από τον πρόεδρο Τραμπ για το αντίστοιχο θέμα. Και στη συνέχεια όχι μόνο έκαναν όλα αυτά, αλλά καθόρισαν ένα πρόγραμμα εργασίας μεταξύ αρχών, ε, πολιτικής προστασίας, κλάδου ε, και ε, φτάνει μέχρι το 2023. Σε ένα από τα έγγραφα που σας έχουμε αποστείλει υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Πότε θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιο είναι το πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει τεχνητά ή φυσικά ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Αντιθέτω, έναντι όλων αυτών των μέτρων, των προληπτικών μέτρων που μόλι σα συνόψα και φτάνουν στο τρίτο σημείο, το αίτημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναφορά μα ε, δεν αναφέρεται καθόλου πουθενά το τεχνητό σκέλος. Αναφερόμαστε μόνο σε φυσική ηλιακή ηλεκτρονομαγνητική ε, ε, ακτινοβολία. Κάτι λείπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να λείπει. Οι μεγάλε καταστροφέ συμβαίνουν από τέτοια πράγματα. Οι μεγάλες καταστροφέ δεν ξεκινούν από την αρχή τη καταστροφή, ξεκινούν ε, μια μέρα σαν τη σημερινή όταν κάποιο πολιτικό δεν έτεινε ε, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δεν έλαβε για υπόψη τι εκκλήσει των οργανώσεων τη πολιτική προστασία, δεν έκαναν κάτι. Επαναλαμβάνω, οι Ηνωμένε Πολιτείε από το 2001 εργάζονται γι' αυτό. Πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρο. Η απειλή είναι τύπου που δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και το ποσοστό είναι πολύ σημαντικό. Θα περάσω απευθεία ε, στο επόμενο σημείο. Δέκα δευτερόλεπτα. Να συνοψίσω τι ζητάμε. Ζητάμε πέντε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που βλέπετε στο χάρτη είναι το σενάριο της τεχνητής ε, ηλεκτρομαγνητικής επίθεσης που το έχει κάνει κάποιος από την Επιτροπή. Είναι επίθεση ε, μιας τρομοκρατικής οργάνωσης με ένα πυρηνικό όπλο το οποίο θα χτυπήσει πέντε ε, ταυτόχρονα διαφορετικές χώρες. Είναι τεράστια η ακτίνα, χιλιόμετρων. Ζητάμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, να δοθεί όθηση για το καθορισμό της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαστημικά φαινόμενα και τη ηλεκτρονομική ακτινοβολία, να υπάρχουν ε, θέματα προστασίας για τους πυρηνικού σταθμού που δεν προστατεύονται. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν ότι πρέπει να καθυστερείτε. Έχουμε την αναφορά σας όλα τα μέλη και επομένως αν θέλετε θα περάσουμε εδώ στις παρεμβάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να ε, σταματήσετε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, δύο πολύ συγκεκριμένα, για τρία δευτερόλεπτα. Θα θέλαμε να ζητήσουμε να συμπεριληφθεί αυτή η απειλή στο πρόγραμμα, να ζητήσουν ε, από, τις, από τα Ηνωμένα Έθνη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μία συνθήκη για τα όπλα αυτά, ε, και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριση αυτών των όπλων ως μηχανισμό πρόληψης και πέμπτον ή δυνατόν να δηλώσουμε την 1η Σεπτεμβρίου ως επέτειο ε, και Ευρωπαϊκή ημέρα για το διαστημικά καιρικά φαινόμενα και την ηλεκτρονική μαγνητική πυροβολία για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Να δω... Ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Λεγκρινιέ έχει το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται πλήρως ε, τις καταστροφικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαστημική μετεωρολογία και στις ε, διαστημικές ε, και πήγες υποδομές αλλά και στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η διαστημική στρατηγική του 2016 καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της αναθεώρησης των διαστημικών προγραμμάτων. Σήμερα έχουμε μια νέα πρόταση κανονισμού που θεσπίζει το νέο διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης. Στον κανονισμό αυτό που είναι υποδιαπραγμάτευση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια νέα συνιστόσα προτείνει ώστε να υπάρχει επιτήρηση του διαστήματος. Ε, συγκεκριμένα μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση για να δούμε ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις ε, που τότε του διαστήματος, ε, σύγκρουση ε, δορυφόρων και κάποιων άλλων, ε, όπως τα λέμε, διαστημικών σκουπιδιών και Και περιμένουμε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένε υπηρεσίες στο πλαίσιο διαστημικής μετεωρολογίας. Θέλουμε δεν να εστιάσουμε σε τιμοπαράδοτες για τους χρήστες, για τους καταναλωτές υπηρεσίες. Για να τις υλοποιήσουμε θα συνεργαστούμε με τους φορείς, τους αρμόδιους. Ήδη έχουν αναπτυχθεί διάφορα έργα και project. Έχουμε το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, για παράδειγμα, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Επομένως, μπορούμε να βασιστούμε στο έργο και στην έρευνα που είναι ήδη στη διάθεσή μας, ώστε να διαθέσουμε σύντομα υπηρεσίες διαστημικής μετεωρολογίας που θα είναι χρήσιμες για τους καταναλωτές. Θέλουμε μια πανευρωπαϊκή διαδικασία για να μπορούμε να αντιδράσουμε όταν έχουμε ένα μείζον συμβάν ε, στον τομέα τη ε, Διαστημική μετεωρολογία. Αυτό είναι η υποσυζήτηση και αντιμετωπίστε στο πλαίσιο του κανονισμού που ανέφερα και ίσω μπορούν να συμπεριληφθούν δραστηριότητε πολιτική προστασία, προστασία του πολίτη, που σημαίνει ότι όταν θα επιλεγούν οι σχετικέ υπηρεσίε Διαστημική Μετρολογία, οι αρχέ προστασία του πολίτη, ε, πολιτική προστασία, θα συμμετάσχουν σε αυτέ τι εργασίε. και Ίσως έχουμε και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιδρούν με συντονισμένο τρόπο. Όποια δράση βέβαια ε, συντονισμού των δράσεων των αρχών πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Αυτά λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό, τα άρθρα που αφορούν την εθνική μετρολογία είναι ένα από τα θέματα ε, επί των οποίων υπάρχει συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, άρα υπάρχει μια κοινή προσέγγιση ήδη από τη 13η Μαρτίου, που σημαίνει ότι οι συνομοθέτες, προς το παρόν τουλάχιστον, επικυρώνουν την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μια τελευταία παρατήρηση πρέπει παρόλα αυτά να σημειώσουμε ότι οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο τη διαστημική Μετρολογία ε, θα είναι περιορισμένου βεληνικού λόγω του προπολογισμού που έχει προταθεί για αυτή την συνιστόσα επιτήρηση του διαστήματος. Πάντως, ε, σίγουρα, τουλάχιστον θα έχουμε ασχοληθεί με αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα και θα μπορέσουμε στο μέλλον να διευρύνουμε τη δράση μα αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ε, θα θέλω τώρα να δώσω το λόγο στους διαφόρους ε, συναδέλφους ε, από το ΕΛΚ καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ροντρίκε Ντία, τον αναφέροντα, για την παρουσία του που μας προειδοποιεί. Προειδοποιεί την Επιτροπή μας για τα ακραία μετρολογικά διαστημικά φαινόμενα και τους κινδύνους που ε, έχουν. Ήταν πολύ διαφωτιστική παρέμβαση, είναι ένα θέμα σημαντικό πολύ σημαντικό, χωρίς ε, να ε, μιλήσουμε κινδυνολογώντας. Ε, υπάρχουν προβλήματα για την ασφάλεια των πολιτών και για κάποιες ηλεκτρο, ηλεκτρικές υποδομές και κρίσιμες ή ηλεκτρομαγνητικές υποδομές πήγες ή στο διάστημα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπε ο κύριος Ρωτήγκεθαρίας. Συμφωνώ και με τις ανησυχίες του και ναι πράγματι πετούνται περαιτέρω προσπάθειες για να γίνουν αντιληφθείς και να διχειριστούμε καλύτερα αυτά τα φαινόμενα, αφού τα γνωρίσουμε καλύτερα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την έρευνα και την ε, καινοτομία σε αυτό το τομέα και έχει ήδη χρηματοδοτήσει καμιά δεκαριά project μαντελοποίησης ε, και πρόβλεψης. Το Μάρτιο, δε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε ένα διαγωνισμό, μια διαγωνισμού. Ε, θέλουμε να ενημερωθούμε για τα έργα τα οποία θα επιλεγούν στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, έχουμε το πρόγραμμα το διαστημικό που θα δώσει απαντήσεις στους κινδύνους που ενέχει η διαστημική μετρόλη και όταν εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει γρήγορα να επιλέξει κομισιόν τις επιχειρησιακές υπηρεσίε ε, διαστημικής μετεωρολογίας και του προμηθευτέ, λαμβάνοντα υπόψη τα ανάγκε των χρηστών. Ο κανονισμός βέβαια ακόμα δεν έχει εγκριθεί, γι' αυτό προτείνω στην Επιτροπή μας να διατηρήσει ανοιχτή την αναφορά και ζητούμε από την Κομισιόν να μας τηρεί ενήμερους για οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Si les parece, como vamos dentro de tiempo y no hay más palabras. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και δεν ε, έχουν ζητήσει το λόγο άλλοι βουλευτές και αυτό θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον αναφέροντα, τον κύριο Ροντρίγε, γιατί τον έκοψα προηγουμένως. Απλά θεωρώ ότι είναι δίκαιο να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο, αλλά αφού δεν υπάρχουν πλέον άλλοι ομιλητές και έχουμε λίγο χρόνο, μπορείτε για 4-5 λεπτά να Μιλήστε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, εμείς είμαστε μια οργάνωση προστασίας του πολίτη. Για 10 χρόνια δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το τομέα, 10 χρόνια και η, ε, το διάστημα μας απασχολεί. Είμαστε 20 χρόνια πίσω και το, λέμε γιατί ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες ε, της μετολογική ε, επιτήρησης ή επίβλεψης 10, μια εβδομάδα μας προστατεύουν. Αν γίνει κάτι Μέχρι να το ε, αντιληφθούμε, έχουμε χάσει το 35%, όπως λένε εκθέσεις του 12, 13, 15, 17. Από 5 έως 50% δεν ξέρουμε ε, δεν έχουμε δυνατότητες. Έχουμε από την άσα ε, ένα ποσοστό 12%. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια απειλή και 1% να είναι η πιθανότητα να υπάρξει, πρέπει να δράσουμε. Τα τελευταία 6 μήνες ε, μια ειδική task force ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εγκρίνει μελέτες ε, από τον Νοέμβριο του 18 και από τον Αύγουστο του 19, δηλαδή πριν από 10 μέρες. Και τις έχετε και τις δύο αυτές Μελέτε τη στείλαμε στη γραμματεία. Αυτή την πρώτη μελέτη λέει ότι αν έχουμε φαινόμενο τέτοιο, 18 ώρες αργότερα θα μας χτυπήσει, όπως έγινε 160 ε, χρόνια πριν, ε, αλλά αυτά γίνονται τα φαινόμενα κάθε αιώνα. Αν γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να έχουμε σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα 99 των αριθμών στην Ανατολική Όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν υπάρχουν πρωτόκολλα προστασία. Και αυτό το λέει μια έκθεση. Και άλλη μια έκθεση στη σελίδα 9 και στη δεύτερη έκθεση του Νοεμβρίου 18, 53 κλπ. στην έκθεση του Αυγούστου 19. Και υπάρχει και μια επιτροπή στη ΣΥΠΑ που αναγνωρίζει ε, ότι θα πρέπει να έχουμε αυτά τα αποθέματα, αποθέματα diesel. Εφτά ημέρες κρατάνε αυτή τη στιγμή για τις αντιδραστήρες. Ε, αν δηλαδή υπάρξει blackout, που μπορεί να κρατάνε και μήνες αυτά τα blackout, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Ε, που είναι 7 μέρες, παραλαμβάνω, μόνο η δυναμικότητα λόγω των αποθέματων που υπάρχουν. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αν υπάρχει πυρκαγιά, αν υπάρξει σεισμό. Πάνω από 130 είναι οι πυρηνικοί αντιδραστήρε και μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη και δεν ξέρουμε πώ θα αντιδράσουν αν υπάρξει ακραίο ε, φυσικό ή τεχνητό ηλεκτρομαγνητικό συμβάν. Γιατί αν πάψουν να λειτουργούν, ε, αν είναι ασφαλή τα εργοστάσια και συνεχίσουν να λειτουργούν, θα μπορούν να είναι μια λύση και να παρέχουν ρεύμα και ενέργεια, αλλά ε, αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Αν σταματήσουν να λειτουργούν δεν θα έχουν ε, αυτονομία πάνω από κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Ε, να μην ε, ψευδόμεθα και να λέμε στον κόσμο, προσπαθώντα να τον καθισχάσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι αυτό ψέμα και το ξέρουμε. Εμεί χρόνια εργαζόμαστε. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό αυτό. Αν γίνει κάτι, 18 ώρες θα μας μένουν και δεν θα έχουμε χρόνο. Στο Rescue, στο Rescue EU, θελήσαμε να υπάρξει και αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή στις άλλε απειλέ ραδιολογικού, χημικού κτλ. πολέμου να περιληφθούν και τα αίτια σε συμβάντα. Δεν περιελήφθη. Θα έχουμε όχι δεκάδες ε, ε θύματα, θα έχουμε εκατόμβε πραγματικά, χιλιάδε θύματα με ένα τέτοιο φαινόμενο, πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς ζητάμε να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με λογικό τρόπο, αντίστοιχα σε αναλογικό τρόπο με αυτά που κάνουν οι Ηνωμένε πολιτείε. Ζητάμε δηλαδή εθνική στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική, όπω αυτή που έχει χαράξει εδώ και τέσσερα χρόνια η Αμερική. Να υπάρξουν μέτρα. Το μόνο που μα ενδιαφέρει είναι αυτό, να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Αν γίνει επίθεση τρομοκρατική, γιατί υπάρχουν διάφορε τρομοκρατικέ ομάδε που προσπαθούν να πάρουν πυρηνικά όπλα στα χέρια του, αυτό είναι μια άλλη ακόμη τεχνητή ε, συνιστώση. Αν έχουμε λοιπόν ε, πυρηνικά όπλα, δεν θα τα βάλουν σε ένα φορτηγό για να προσπαθήσουν να καταστρέψουν ε, μια πόλη, αλλά από μια βάρκα, από ένα πλοίο μέσα σε διεθνή ύδατα, στα 200 μίλια για παράδειγμα, αν το βάλουν σε έναν εκτοξευτήρα, μπορούν να δημιουργήσουν εθνικό blackout με τρομερές επιπτώσεις σε ε, για τις οποίες δεν είμαστε προετοιμασμένοι σήμερα. Λένε κάποιοι ότι δεν είναι του σήμερα κάτι τέτοιο. Όχι. Ε, ισχύει και πρέπει να το ξέρουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι. Να διαβάσετε τα έγγραφα. Είπανε όλα επίσημα. Επίσημε με τελευταία πριν 10 ημέρε, όπω σα είπα, μελέτη. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και εσεί που παίρνετε τι πολιτικέ αποφάσει πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τα αναφέροντα, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούσαμε και την ε, βουλευτή, οπότε πρόταση είναι να μια ανοιχτή αναφορά για να συνεχίσουμε να εξετάζουμε και να μελετούμε το θέμα. Ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουμε αυτός ο κανονισμός ε, για το διάστημα να εγκριθεί, ώστε να παληθεύσουμε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό είναι επαρκής και κατάλληλη. Και επίση ζητούμε να μα στηρεί ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλε τι πρωτοβουλίε στον τομέα αυτό, τον τόσο σημαντικό. Να τηρείτε λοιπόν ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακαλούμε. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση την αναφορά αυτή, ολοκληρώνεται και η συνεδρίασή μας για σήμερα το πρωί και θα τα ξαναπούμε στις 2.30 το μεσημέρι για να δούμε τις υπόλοιπε αναφορές μερίσιας διάταξης. Αριστούμε και ιδίως τον αναφέροντα.